Και δίνω λοιπόν το λόγο στον Επιτρόπο Δήμα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρος. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε εκείνους που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Φέτος το καλοκαίρι η κοινότητα είχε σημαντική συνεισφορά στην κατάσβεση των πολλών και δύσκολων δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε διάφορα κράτη μέλη. το πιλωτικό πρόγραμμα της τακτικής ευρωπαϊκής εφεδρείας πυρόσβεσης της ευρωπαϊκής ένωσης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και παρήχε βοήθεια στα κράτη μέλη που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές. θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που ενέκρινε τη χρηματοδότηση του πιλωτικού αυτού προγράμματος. Πρέπει να πω επίσης ότι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα είναι μέρος, μικρό μέρος, είναι υλοποίηση των προτάσεων και ιδεών ε, της έκθεσης Μπαρνιέ, του Μισελ Μπαρνιέ, στον οποίο επίσης εκφράζω την, ε, τις ευχαριστίες μου. Με αυτό το πιλωτικό ε, πρόγραμμα ενισχύθηκε ουσιαστικά ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας και κατά συνέπεια η δυνατότητα συνεισφοράς ε, σε χώρες ε, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης προσέφεραν εναέρια μέσα πυρόσβεσης στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες. Για πρώτη φορά μάλιστα δύο κοινοτικά πυροσβεστικά αεροσκάφη συμμετείχαν μαζί με τα ελληνικά με τα πορτογαλικά με τα γαλλικά εναέρια μέσα στην προσπάθεια κατάσβεσης στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος για τη δημιουργία αυτόνομης κοινοτικής δύναμης πυρόσβεσης με αφορμή αυτέ τι ε, πυρκαγιέ, τι πρόσφατες πυρκαγιές πολλές ήταν πάλι φωνέ φωνές που ακούστηκαν από πολιτικού, επιστήμονε, δημοσιογράφου, απλού πολίτε για την ανάγκη δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια εξειδικευμένη δύναμη αντιμετώπιση πυρκαγιών η οποία να μπορεί να επεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά όταν τα εθνικά μέσα πυρόσβεσης δεν επαρκούν. Ε, έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή Προ τη δημιουργία δηλαδή μια αυτόνομη δύναμη επέμβαση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και ε, όπω είπα η συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν καθοριστική. Μα επέτρεψε να εξασφαλίσουμε κονδύλια για την ενοικίαση πυροσβεστικών αεροσκαφών και για πρώτη φορά φέτο, το καλοκαίρι συστήσαμε και θέσαμε σε λειτουργία από την περίοδο από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δύναμη αεροπυρόσβεση υπό την εποπτεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ευρωπαϊκή Τακτική Εφεδρεία δασοπυρόσβεση αεροσκάφη τη οποία συμμετείχαν στι επιχειρήσεις πυρόσβεση ε, στι ε, διάφορες χώρες, συγκεκριμένα σε έξι περιπτώσεις από τις εννέα στις οποίες εκλήθη ο μηχανισμός ε, πολιτικής προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωση, για τον οποίο κινητοποιήθησαν. Πράγματι ανάμεσα στα εθνικά είτε ελληνικά είτε πορτογαλέζικα είτε ιταλικά εναέρια μέσα ε, και σε αυτά τα οποία ήρθαν από άλλες χώρες συμμετείχαν και τα αμυγός κοινοτικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία μάλιστα επιχειρούσαν με τα διακριτικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι κάποιου κράτους μέλους. Το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα έχει σαν στόχο να καλύψει τυχόν κενά στο εναέριο δυναμικό των κρατών μελών και όχι να υποκαταστήσει τα διαθέσιμα εθνικά μέσα τα αναβλωμένα εφεδρικά αεροσκάφη χρησιμοποίησαν φέτος ε, όπως είπα στην πορτογαλία στην νότιο γαλλία και κορσική στην ιταλία και στην ελλάδα ε, στην περιοχή της αττικής όπου είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές. Ε, εδρεύουν στην νήσο κορσική η οποία βρίσκεται σε ίση απόσταση επέμβαση από τα δύο γεωγραφικά άκρα της μεσογείου. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θεωρώ ότι είναι επίγουσα πλέον η ανάγκη αυτόνομη ικανότητα σε αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε κοινοτικό επίπεδο. ελπίζουμε ότι το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα θα αποτελέσει τον πυρήνα μια μελλοντική ευρωπαϊκή δύναμη, ταχεία επέμβαση και καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών ε, ή και άλλων ε, φυσικών ε, καταστροφών ή καταστροφών που προκαλούνται από τον άνθρωπο. βεβαίω υπάρχουν ορισμένε διαφορετικέ. Ε, σκέψεις σχετικά ειδικότερα για το θέμα των δασικών πυρκαγιών. Ε, ορισμένοι επικαλούνται την αρχή της επικουρικότητας στον τομέα της διαχείρισης και της προστασίας του δασικού πλούτου. Ε, επίσης υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς την παραχώρηση περαιτέρω αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Επίσης υπάρχουν επιχειρήματα ότι η ύπαρξη μιας ευρωπαϊκής δύναμης αντιμετώπισης πυρκαγιών θα έδινε μια πλαστή αίσθηση ασφάλειας σε πολλές εθνικές αρχές οι οποίες ενδεχομένως θα παραμελούσαν τις απαραίτητες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό σε μέσα καταπολέμησης και κυρίως στον τομέα της πρόληψης των πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών. πέρα από αυτές τις ε, αντιδράσεις ε, προκύπτουν και ορισμένα πρακτικά προβλήματα ε, προβλήματα συντονισμού ειδικότερα για το θέμα των δασικών πυρκαγιών με βάση ποια κριτήρια και ποιες προτεραιότητες θα καθορίζονται και πώς θα χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκές Αναέριες μονάδες πυρόσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές χώρες ταυτόχρονα παραδείγματος χάρη στην πορτογαλία και στην ελλάδα ταυτόχρονα. όλα αυτά τα ζητήματα πάντως θα αναλυθούν σε έκθεση που θα υποβάλει η ευρωπαϊκή επιτροπή προς συζήτηση στο συμβούλιο υπουργών ε, και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αναφορικά με τη λειτουργία του πολιτικού προγράμματος ε, του πιλωτικού προγράμματος το φετινό καλοκαίρι. Ε, πρέπει ε, και το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο ε, να πιστούν και η Επιτροπή και να συνεργαστούν για την δημιουργία αυτού του μηχανισμού. Βεβαίως, ενδιαμέσως, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μην αμελούν ούτε στο ελάχιστο τις υποχρεώσεις τους στον τομέα της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της πρόληψης. θα πω δύο κουβέντες ακόμη για το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 2001 και ο οποίος ε, τα πρώτα έτη ε, λειτουργούσε ε, με λίγες παρεμβάσεις. Από το 2005 και μετά έχουμε υπερπολαπλασιάσει, πενταπλασιάσει τις επεμβάσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 50% εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, 50% εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ το συντονισμό αλλά και την βοήθεια την οποία ε, παρέχουμε μέσω του μηχανισμού ε, τη ε, πολιτική προστασία. Και είναι γνωστό πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση τόσο στο, στην περίπτωση του τσουνάμι όσο και στην κατρίνα. Μάλιστα και στις δύο αυτές τις περιπτώσεις ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι οι οποίοι στείλαμε ε, ειδικού ε, στους ε, τόπους των καταστροφών. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως έχουμε πολλά να κάνουμε και όποιος διαβάσει την έκθεση Μπαρνιέ θα δει πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε τον, την πολιτική προστασία επόφελος των Ευρωπαίων πολιτών και την προστασία βεβαίως του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε Δήμα. Και περνάμε τώρα ε, στη συζήτηση εκ μέρου των ε, ομάδων. Ο κ. Κυλακάκης, εκ μέρου του ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Νότια Ευρώπη καταστρέφονται κάθε χρόνο 400.000 εκτάρια δασών. Πρόκειται για μια καταστροφή μεγάλου μεγέθους και συστηματικότητας στις επόμενες δεκαετίες το πρόβλημα θα χειροτερέψει. για 30 με 40 χρόνια τουλάχιστον θα ζήσουμε ό,τι και να κάνουμε από πλευράς μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου μια επιδείνωση, μια κλιματική επιδείνωση η οποία ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη όπου τα δάση είναι ευάλωτα θα την βιώσουμε αρνητικά θα ζήσουμε στο μέλλον περισσότερο μεγάλες πυρκαγιές και χειρότερους κινδύνους. Υπό κανονικές συνθήκες η αντιμετώπιση των πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα και υποχρέωση των κρατών μελών. Και τα κράτη-μέλη στην Νότια Ευρώπη αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες πυρκαγιές το χρόνο με επιτυχία. Κάθε τόσο όμως υπό εξαιρετικές συνθήκες υπάρχουν πυρκαγιές μεγάλης καταστροφικότητας όπου η εξωτερική βοήθεια και αλληλεγγύη είναι αναγκαία. το σχέδιο απόφασης που προτείνουμε εκ μέρους του ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος στηρίζεται σε αυτές τις διαπιστώσεις και αναδεικνύει μεταξύ άλλων πόσο επίγουσα είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής δύναμης άμεσης επέμβασης στην οποία αναφέρθηκε ο επίτροπος κ. δήμας και η οποία προτείνεται στην έκθεση Μπαρνιέ. την ανάγκη ευέλικτης και άμεσης κινητοποίησης των πόρων του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλεγγύης την ανάγκη να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα οι δασικές πυρκαγιές στη νότια ευρώπη στο επεξεργασία σχέδιο δράσης της ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή την ανάγκη να υποβληθεί το ταχύτερο η πρόταση της επιτροπής για μια ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. για τη χώρα μου και προφανώς για τους πολίτες που επλήγησαν είναι σημαντικό η απόφαση αυτή να υπερψηφιστεί από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. είναι σημαντικό το σώμα να δείξει την ευαισθησία του σε αυτό το κρίσιμο για την νότια ευρώπη θέμα. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Ποδηματά, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Φέτος, για μια ακόμη χρονιά, η ιστορία των δασικών πυρκαγιών επαναλαμβάνεται επιδεινώνεται και ερχόμαστε κάθε φθινόπωρο κατόπιν εορτής να συζητήσουμε για την αποκατάσταση των πληγυσών περιοχών και την ανακούφιση των πληγέντων. στην ελλάδα θρηνούμε και πάλι φέτος εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια καμένης γης ανυπολόγιστης οικολογικής και οικονομικής καταστροφής ενώ αντίστοιχη είναι η έκταση της καταστροφής και στην ισπανία την πορτογαλία την ιταλία και τη γαλλία ένα πράγμα κύριε επίτροπε είναι σαφές και το υπενηχθήκατε ότι δεν καταφέρνουμε να αντλήσουμε μαθήματα από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος. εδώ και έξι τουλάχιστον χρόνια μιλάμε για μια κοινή ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας πάγιο αίτημα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της οποίας όμως η σημασία απαξιώνεται από τα λάθη ορισμένων εθνικών κυβερνήσεων λάθη στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή αποτρεπτικών μηχανισμών και μέτρων πρόληψης αδυναμία ή αβουλία επιβολής αυστηρής νομοθεσίας που να καθιστά υποχρεωτική την αναδάσωση των κατεστραμμένων περιοχών μη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων για την αποκατάσταση των πληγέντων. στο κοινοτικό επίπεδο πέρα από τη δύναμη πολιτικής προστασίας η άμεση ενεργοποίηση των κονδυλίων του ταμείου αλληλεγγύης και κυρίως η αποδέσμευσή του από τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς οφείλουν να αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της επιτροπής. τέλος κύριε επίτροπε γνωρίζετε καλά καλύτερα από εμάς ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα γενιά πυρκαγιών τις λεγόμενες πυρκαγιές υψηλής έντασης οι οποίες συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και πλήττουν κυρίως τα δάση της μεσογείου και της νότιας ευρώπης χρειαζόμαστε λοιπόν άμεσα επανασχεδιασμό της δασικής προστασίας σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο με προσαρμογή της πρόληψης και της αντιμετώπισης πυρκαγιών στα νέα δεδομένα και ένταξη των πολιτικών αυτών στο πλαίσιο των δρομολογούμενων μέτρων για την προσαρμογή των χωρών μελών στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους και δημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Μπιλμπάου, 1,5 λεπτό. Κυρία Μπιλμπάου, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τον Επιτροπό για τις εξηγήσεις. Πράγματι πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινοτική πολιτική ε, στα θέματα πρόληψης. Πρώτα απ' όλα ε, όσον αφορά ε, τις φωτιές αυτές, πυρκαγιές αυτές που είδαμε να έχουν ξεσπάσει σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ξεκινώ την παρέμβασή μου υπενθυμίζοντας τους τέσσερις αυτούς πυροσβέστες που πέθαναν τον περασμένο Ιούλιο στην Ταραγώνα και να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μας προς, όλες, προς τις οικογένειές Σημαντική η πολιτική πρόληψη αλλά και σημαντική η πολιτική συντονισμού. Μην ξεχνάμε ότι πολλέ από τι ε, πυρκαγιέ που ξέσπασαν ε, συνδέονται ε, γύρω από κερδοσκοπικέ δραστηριότητε, Από... Υπάρχει υπόνοια δηλαδή ότι έγιναν για, για λόγους άλλους, για πολυδομικούς σκοπού. Πρέπει λοιπόν να, είναι πιο, να υπάρξουν πιο αυστηρέ ποινέ για αυτά τα αδικήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Και επίση πρέπει πρέπει να μελετήσουμε ε, και την δίωξη μέσω ευρωπαϊκού Εντάλματο. Πρέπει ταυτόχρονα να δοθούν οι απαραίτητοι πόροι έτσι ώστε να αναπτυχθούν μηχανισμοί καινοτόμοι έτσι ώστε να μπορεί να γίνονται σωστά και με ακρίβεια η μέτρηση του ανέμου, ε, της θερμοκρασίας, έτσι ώστε ε, σε επίπεδο πρόληψης να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Για τους πράσινους, ο κύριος Τρεμόπουλος. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πράγματι ενδιαφέρον το ότι κυρίως οι Έλληνες μιλούν για αυτό το τεράστιο θέμα που απασχολεί όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο μια και καταστρέφονται τακτικά από τεράστιες δασικές πυρκαγιές μεγάλες εκτάσεις και υποβαθμίζουν ε, την ποιότητα ζωής τη βιοποικιλότητα την περιφερειακή ανάπτυξη και το μέλλον των πολιτών συχνά οι δασικές πυρκαγιές όπως ε, πρόσφατα στην ε, ελλάδα οφείλονται σε ελλειπείς και αντικρουόμενες δασικές και οικιστικές πολιτικές που ευνοούν τους εμπρισμούς και τις παράνομες ενέργειες με στόχο την εκποίηση των δασικών εκτάσεων. δυστυχώς και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν προσπαθήσει να αμβλύνουν να μειώσουν τη συνταγματική προστασία των δασών οι συνεχείς πιέσεις για αλλαγή των χρήσεων γης και για επέκταση των οικισμών και βέβαια οι ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι που καίγονται ή και αυτοαναφλέγονται σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή που για κάποιους είναι απλά άλοθη αυξάνουν πια τις πιθανότητες για περισσότερες φυσικές καταστροφές. είναι λοιπόν σημαντικό να εστιάσουμε περισσότερο στην πρόληψη την προστασία και την έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από συντονισμένε και συνεργατικέ δράσει. σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή μιας κοινή ευρωπαϊκής βιώσιμης πολιτικής για τα δάση και να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα από τα ταμεία συνοχή της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης που προορίζονται για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καθώς και για την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών χρησιμοποιούνται όντως με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο. τα κονδύλια που δίνονται για την αποκατάσταση των ε, πληγέντων περιοχών πρέπει να αξιοποιούνται στη βάση ορθολογικών μέτρων αναδάσωσης αλλά και επιστημονικών μελετών ενώ τονίζουμε ότι πρέπει να επιστρέφονται από τα κράτη μέλη όταν διαπιστώνεται ο αποχαρακτηρισμός των πληγέντων δασικών εκτάσεων προς όφελος της οικιστικής ή της τουριστικής ανάπτυξης. στο παρελθόν και μόλις πριν από δύο χρόνια το κοινοβούλιο έχει κάνει συστάσεις με ψηφίσματα για την πρόληψη και την κέρια αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων που δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο πιστεύουμε ότι η μακροχρόνια προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας είναι εφικτή μόνο μέσα από την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών τη συγκράτηση του πληθυσμού των ε, ανθρώπων της υπαίθρου και τη δημιουργία νέων πράσινων επαγγελμάτων την διαβίω εκπαίδευση και κατάρτιση την ενδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών με έμφαση στις εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης. τέλος πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μηχανισμών έγκαιρης αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών μέσα από την ενδυνάμωση της μόνιμης δύναμης πολιτικής προστασίας που ανέφερε ο κύριος δήμας αλλά και την παραπέρα αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αναφοράς μπαρνιέ. σε αυτά τα πλαίσια καταθέτουμε ψήφισμα σήμερα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με την ελπίδα ότι θα κάνουμε κάποιο βήμα σε ό,τι αφορά τη σύμπραξη και τη συνεργασία των κρατών για μια ουσιαστική πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών αλλά και την πιο αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ευρωπαϊκής ένωσης για τον σκοπό αυτό. το χρωστάμε στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χουντής. από την Γκουε για 1,5 λεπτό. Ελπίζω σωστά να προφέρω το όνομά σας. Η χώρα μου, η Ελλάδα, για τρίτη συνεχή χρονιά βιώνει τεράστια έκταση καταστροφικές πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές του 2007, από τις χειρότερες τραγωδίες αυτού του είδους, αλλά και οι φετινές στη βορειοανατολική Αττική, ανέδειξαν τη γύμνια του συστήματος αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας. Θυμίζω ότι η Ελλάδα, η Αθήνα, συγγνώμη, είναι η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που έχει τη μικρότερη αναλογία σε πράσινο ανακάτοικο που έχει τους υψηλότερους ατμοσφαιρικούς ρήπους και οι πυρκαγιές του 2007 και του 2009 έχουν επιδεινώσει το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μπορεί οι κλιματολογικές αλλαγές να ερμηνεύουν ως ένα βαθμό τις καταστροφές που έχουμε στη νότια Ευρώπη. Όμως υπάρχουν ελλείψεις και στις εθνικές πολιτικές και στην πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης στο βαθμό που δεν έχει ενσωματώσει ικανοποιητικά την κλιματική αλλαγή στην περιβαλλοντική στρατηγική. οι ελληνικές κυβερνήσεις ανέχονται να δομούνται καμένες περιοχές και να σφετερίζεται η δημόσια περιουσία ενώ υπάρχει ανελαστικότητα από τα ταμεία της ευρωπαϊκής ένωσης. κατόπιν τούτου κύριε επίτροπε κύριε δήμα θέλω να σας ρωτήσω προτίθεται η ευρωπαϊκή επιτροπή να συμβάλει στη θεσμική θωράκιση των δασών της χώρας με την άμεση κινητοποίηση της διαδικασίας κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών που αν υπήρχαν ίσως είχαμε αποφύγει αυτούς τους εμπρισμού. προτίθεται να συγχρηματοδοτήσει άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα προκειμένου να μην υπάρξουν νέες καταστροφές στις πληγείσες περιοχές; προτίθεται να προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις των κατάλληλων αναδασώσεων διότι δεν γίνονται σε επαρκή αναπλήρωση των καταστροφών; και τέλος προτίθεται η ευρωπαϊκή επιτροπή να, συζητήσει με την όποια νέα κυβέρνηση προκύψει από τις ε, ε, επόμενες εκλογές στην ελλάδα για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στο πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού που θα δώσει ανάσα ζωή στην αττική. Σα ευχαριστώ πολύ και εύχομαι χρόνια πολλά για την ονομαστική γιορτή του κυρίου επίτροπου όπω λέμε στην ελλάδα. Ευρώπης, η κυρία Τζαβέλα, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, πολύ χάρηκα που σας είδα και σας άκουσα. Ε, θεωρώ ότι αυτά που είπατε ήταν και η απάντηση στην επιστολή που σας στείλαμε τη δεύτερη μέρα των πυρκαγιών, όπου είχαμε την πρόταση για μια κοινή δράση του Νότου της Ευρώπης όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και συγκεκριμένες προτάσεις εξειδικευμένες που σας είχαμε κάνει. Επίσης θέλω να πω κύριε Επίτροπε ότι πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι όλοι οι άλλοι ευρωβουλευτές των ελληνικών κομμάτων και του Ισπανικού κόμματο ανταποκριθήκαν στην έκκληση που κάναμε για μια κοινή παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο και κοινή προσπάθεια για τη χάραξη μιας ε, ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Κύριε Επίτροπε, από ό,τι φαίνεται οι κλιματικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Οι κλιματικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο δομικό φαινόμενο πλέον. Είναι δομικό φαινόμενο οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, τις οποίες παρατηρούμε μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε. Θα έπρεπε κύριε Επίτροπε να θέσουμε τις ε, βάσεις για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενωθούν οι κυβερνήσεις των μεσογειακών κρατών σε μια προσπάθεια να πείσουν τους βόρειους εταίρους μας για την αναγκαιότητα αυτού του μηχανισμού που είπατε τόσο στα πλαίσια της επικουρικότητας όσο και στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Κατάλαβα κύριε Επίτροπε ότι έχετε προβλήματα όσον αφορά τον, την τήρηση της επικουρικότητας από τη Βόρεια Ευρώπη. Εύχομαι το φαινόμενο των φυσικών καταστροφών να είναι μόνο στη νότια ευρώπη. πολύ φοβάμαι όμως ότι οι κλιματικές αλλαγές προχωρούν με τόσο μεγάλη ταχύτητα που μπορεί να έχουμε φυσικές, αλλαγές, ε, καταστροφές άλλου χαρακτήρα και στη βόρεια ευρώπη. πολύ καλά λοιπόν κάνετε και προτείνετε προληπτικά να χαράξουμε αυτή τη στρατηγική της ε, πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών ε, φαινομένων. προς το παρόν υπάρχει αυτή η μικρή μονάδα που εδρεύει στην Κορσική. Λειτουργήσε καλά το καλοκαίρι, είναι επιτακτική ανάγκη αυτή η μονάδα να αναπτυχθεί και να στηριχθεί ο Επίτροπος Περιβάλλοντος στη σχετική με το θέμα εισήγησή του τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο και θα έκανε έκκληση προς τους ευρωβουλευτές των χωρών του Νότου να συνεργαστούν με τις ε, κυβερνήσεις τους και να στηρίξουν τις εισηγήσεις του κυρίου Δήμα και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, το οποίο είναι προς όφελος όλων των χωρών του Νότου. Ε, είδα την ε, πρόταση του ΕΛΚ και πράγματι με βρίσκει σύμφωνη. Ε, θα προσέθετα και χαίρομαι πράγματι που προχωρήσανε αυτό το ψήφισμα θα προσέθετα και κάτι άλλο σε αυτό το ψήφισμα το οποίο προωθεί το ελκ έχοντας ως αρχή ότι οι κλιματικές αλλαγές ήδη έχουν ως αποτέλεσμα τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες στη διάσκεψη της κοπενχάγης θα πρέπει η επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην χάραξη στρατηγικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών να ορίσει προϋπολογισμό που θα χρειαστεί για να καλύψει πρόληψη και καταστολή φυσικών καταστροφών στην Κοπεχάγη να ενισχύσει προς το σκοπό αυτό την πρότυπη μονάδα της Ευρωπαϊκής Τακτικής Εφεδρείας Δασοπυρόσβεσης. Αναμένουμε κύριε Επίτροπε να δούμε στην ατζέντα της Κοπεχάγης πολύ υψηλά και σε πρώτη προτεραιότητα την ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Όμπερμαϊρ για δύο λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αυτά που ζήσαμε στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να επαναληφθούν ποτέ στην Ευρώπη. 75 πύρος ε, φωτιές είχαμε στην Ελλάδα, στα βόρεια της Αθήνας, οι πιο πολλές εξ αυτών ανεξέλεκτες. Και όλα αυτά Και μάλιστα οφείλεται σε ε, θελοντικές δράσεις το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις περιορίστηκε η ανθρώπινη τραγωδία. Οι εθελοντές ε, πυροσβέστες ε, θα πρέπει να τους συγχαρούμε ιδιαίτερα και λέω φίλους και συναδέλφους γιατί και εγώ είμαι εδώ και πολλά χρόνια μέλος της εθελοντικής πυροσβεστικής ε, στην Αυστρία και ξέρω τι προσπάθεια καταβάλλεται. Χωρί τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Να πω για την Επιτροπή το εξή. Ε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό να υπάρχουν κοινοτικέ δυνάμει για να συνδράμουν το εθνικό έργο, όταν δεν αρκούν οι εθνικές ε, δυνάμεις. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί πολιτικής προστασίας και θα πρέπει να συστήσω στο σημείο αυτό να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε προκειμένου για παράδειγμα, στην κεντρική Ευρώπη, στην Γερμανία, στην Αυστρία υπάρχουν εθελοντικά τέτοια συστήματα τα οποία καλύπτουν ε, την περιφέρεια. Και νομίζω, και το συστήνω στους Έλληνες φίλους, ότι είναι ενδιαφέρον να δραστηριοποιείται ο καθένας σε αυτές τις ε, περιπτώσεις και αν στις ε, περιφέρειες αυτές υπάρχει η επιθυμία να συσταθούν τέτοια εθελοντικά προγράμματα, εγώ προσωπικά είμαι πρόθυμος να συνδράμω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτή ήταν οι ομιλητές εκ μέρους των ομάδων και περνάμε τώρα στους περαιτέρω ομιλητές. Ο κύριος Μπαρνιέ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίω θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που είναι παρόν και για τις απαντήσεις που έδωσε και την προσοχή που συνεχίζει να αποδίδει σε όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ μαζί όταν ο πρόεδρος Μπαρόζο μας ζήτησε να συντάξουμε μια έκθεση την οποία ανέφερε για, μια, για τη δημιουργία μιας δύναμης πολιτικής προστασίας ευρωπαϊκής. Την με αυτή την έκθεση το 2006 και όταν την ξαναδιαβάζω και σκέφτομαι και όλες τις καταστροφές που έχουν επέλθει πραγματικά είναι επίκαιρη. Κυρία Τζαβέλα βεβαίω δεν είναι μόνο η Ελλάδα, ενδιαφέρονται πάρα πολλέ χώρες. Δεν υπάρχουν μόνο οι φυσικές καταστροφέ, υπάρχουν και οι ανθρώπινες καταστροφέ που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, ε, το έρικα, ε, τα βιομηχανικά ατυχήματα τύπου Τσερνομπίλ. Υπάρχουν δηλαδή καταστροφές ε, άλλες εκτός από τις πυρκαγιές και φυσικές. Ένα τσουνάμι στη Μεσόγειο μπορεί να επισυμβεί αυτό όπως υπήρξε στην αρχή του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τελικά ε, ε, απόλυτα την πόλη της Μεσίνης. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα εργαλεία, οι μηχανισμοί που κινητοποιούμε δεν ανταποκρίνονται στις καταστροφές οι οποίες πολλαπλασιάζονται κάτω από την υπερθέρμανση του κλίματος και λόγω των μεταφορών. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Δήμα και τις Γενικές Διευθύνσεις που ε, λειτουργήσαν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο με τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενισχυμένη συνεργασία. Ας μην είμαστε 27, ας είμαστε 12 ή 15 και θα δείτε ότι σιγά σιγά θα ενδιαφερθούν όλοι. Όταν κάνω τον κατάλογο των καταστροφών, όλοι ενδιαφέρονται. Πλημμύρες στη Γερμανία το 2002, ε, πανδημίες, τρομοκρατία. Γι' αυτό θα ήθελα η Επιτροπή, κύριε Επίτροπε, να αναλάβει την πρωτοβουλία να ε, προτείνει στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν και το Κοινοβούλιο μας ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην, ε, σε άλλες επιτροπές θα σας υποστηρίξουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Στρέλα για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, κοιτάξτε εδώ για άλλη μια φορά Μιλάμε για τις ε, δασικές πυρκαγιές. Μα κοιτάξτε, κάθε χρόνο οι πυρκαγιές ε, καταστρέφουν μέρος των δασών μας και με τις κλιματικές αλλαγές ε, τα πράγματα δεν ε, φαίνονται περισσότερο βίωνα για το μέλλον. Οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να αποφευχθούν απόλυτα, αλλά βεβαίως πρέπει να προσπαθήσουμε να τις αποφεύγουμε μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου και καθορίζοντας μια σαφή, μια σωστή δασική πολιτική που θα μας επιτρέψει να αναγνωρίσουμε το πόσο σημαντικά είναι τα δάση ε, και τι υπηρεσίες προσφέρουν ε, στο ε, περιβάλλον, κυρίως στον τομέα του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή. Σε πολλά κρατημέλη έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις για την, προ καταπολέμηση των πυρκαγιών. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, εγκρίναμε ένα σχέδιο ε, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα κονδύλια για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Αναθεωρήσαμε την νομοθεσία μα ε, όσον αφορά την αναδάσωση των ε, περιοχών που πλήττονται και παρόλα αυτά εξακολουθούμε να έχουμε πυρκαγιέ. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε περισσότερε προσπάθειε σε όλα τα κρατημέλη που πλήττονται από το φαινόμενο αυτό. Ταυτόχρονα θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει τις προτάσεις που έχει υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορα ψηφίσματα. Υπάρχουν διάφορα έγγραφα τα οποία αναφέρουν συγκεκριμένες λύσεις. Αναφέρθηκε ήδη το έγγραφο Μπαρνιέ. Υπάρχουν και άλλα που έχουν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Και εγώ η ίδια ήμουν συγκήτρια μια έκθεση για τι φυσικέ καταστροφέ στην Επιτροπή Περιβάλλοντο και θα, ε, πρέπει να σας πω ότι έχω κάνει και εγώ μια σειρά προτάσεων. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε στα κράτη-μέλη τα οποία ε, εκφράζουν αντιρρήσεις οικονομικής φύσεως, να πούμε ε, το εξής. Στην ουσία, είναι πολύ πιο δαπανηρό να διορθώνουμε την κατάσταση παρά να προλαμβάνουμε το κακό και λαμβάνοντα υπόψη και τη συνδιάσκεψη τη Κοπεχάγη, χρειαζόμαστε ένα φιλόδοξο σχέδιο για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη και θέλουμε να έχουμε επίτροπε ένα συγκεκριμένο σχέδιο τη πυρκαγιά όπω και τι πλημμύρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φέτος το καλοκαίρι και η Κωσική ήταν θύμα μεγάλων πυρκαγιών όπως η Σαρδινία, η Καταλωνία, η Ελλάδα, η, τα Κανάρια και τόσες άλλες περιοχές της Ευρώπης. Για όλους τους πληθυσμούς που υπέστησαν αυτές τις πυρκαγιές, η ομάδα μας θα ήθελε να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θέτοντας σε κίνηση το Ταμείο το σχετικό. Τι θα κάνει η Κομισιόν λοιπόν σχετικά κύριε Επίτροπο με το Ταμείο Αλληλεγγύης. 23 Ιουλίου φέτος στην Κορσική είχε πάρα πολύ ζέστη 44 βαθμούς, ξερός αέρας, έντονος αέρας και αυτό συμβαίνει όλο και περισσότερο συχνά λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τοπικές δυνάμεις είχαν ε, ξεπεραστεί ενώ πέρυσι τα πράγματα ήταν πιο απαλά και είχε γλιτώσει η Κορσίκη. Το μάθημα για μένα είναι απλό. Όταν υπάρχουν τέτοιες μετρολογικές συνθήκες που προβλέπονται, πρέπει να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ε, Δύναμης Πολιτικής Προστασίας, όπως προβλέπεται στην έκθεση Μπαρνιέ, ώστε να παρέμβουμε προτού επεκταθούν τα πράγματα, διότι αφού η μπει στο δάσος, τότε πρέπει, θα καεί όλο το δάσος. Δεν σταματήσει αλλιώ. Αναφερθήκατε σε ένα πρόγραμμα πιλότο, κύριε Επίτροπε. Θέλουμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν ώστε οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας να ανταποκριθούν το ταχύτερο δυνατόν στην προστασία, για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Μεσόγειο. Δεν είναι φυσικό ο προϋπολογισμός να μην προβλέπει τίποτα το 2010 για αυτές τις δυνάμεις. Υποβάλαμε τροπολογία και το και δέχεται να μας υποστηρίξει για να περάσει αυτή η τροπολογία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τούσας, 1,5 λεπτό. Οι πυρκαγιέ είναι βαθιά πολιτικό πρόβλημα που με ιδιαίτερη οξύτητα παρουσιάζεται στι χώρε όπω είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα με οδυνηρέ συνέπειε σε ό,τι αφορά του λαού αλλά και το περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία μα από την Ελλάδα. Οι πυρκαγιές που κατέκαψαν την βορειοανατολική Αττική τον κιθερώνα την εύβοια και άλλες περιοχές της ελλάδας προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές είναι αποτέλεσμα της εμπρηστικής πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης και των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων και στη χώρα μας που θέλει τη γη τα δάση και τους ορεινούς όγκους εμπόρευμα της καπιταλιστικής οικονομίας. αυτή η άκρος επικίνδυνη πολιτική οπλίζει το χέρι των εμπριστών που σύμφωνα με τα γεγονότα και τις καταγγελίες κατοίκων αυτών των περιοχών που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές και αυτή τη φορά έδρασαν βάσει σχεδίου. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Ο οποιοδήποτε μηχανισμός όσο και αν εξοπλιστεί με το πιο σύγχρονα μέσα εάν δεν αντιμετωπιστούν τα ουσιαστικά προβλήματα της εμπορευματοποίησης και της αλλαγής χρήσης της γης δεν θα μπορέσουμε να ανακόψουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που καταστρέφει το περιβάλλον ε, υποθηκεύει το μέλλον του πλανήτη γενικότερα οι πρώτες τραγικές συνέπειες αυτής της πολιτικής εκδηλώθηκαν ήδη στην εύβοια στις 12 σεπτέμβρη του 2009 πριν από λίγες μέρες με τις καταστροφικές πλημμύρες που έπνιξαν την πυρόπληκτη εύβοια. τα ελλειπή αντιπλημμυρικά έργα και το σαθρό από τις πυρκαγιές έδαφος σε συνδυασμό με την ένταση της βροχής προκάλεσε το θάνατο ενός ατόμου τεράστιες καταστροφές σε χωριά δρόμους γέφυρες και άλλες υποδομές η καταστροφή αυτή δεν δικαιολογείται από τη σφοδρή βροχόπτωση. Δεν είναι μοιραίο σε κάθε φυσικό φαινόμενο. Οι εργαζόμενοι να θρυνούν ζωέ και κατεστραμμένοι περιβάλλον. Είναι επιτακτική ανάγκη να χρηματοδοτηθούν άμεσα μέτρα καταγραφή των ζημιών αποζημίωση των πληγιστών λαϊκών οικογενειών της αγροτιάς και των κτηνοτρόφων καμία αλλαγή χρήσης γης αναδάσωση των καμένων εκτάσεων να μετατραπεί σε δημόσια περιουσία η διοκτησία των μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων στα βουνά και τα δάση και επιπρόσθετα ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των δυνάμεων της δασικής υπηρεσίας ως δημόσιας υπηρεσίας που θα έχει Σας ευχαριστώ. Ακόμα και αν δεν έχουμε χρονική πίεση σήμερα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάπως να τηρούμε τη χρονική, το χρόνο που έχει ο καθένας στη διάθεσή μας. Από σεβασμό προς τους συναδέλφους που τηρούν το χρόνο τους. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μαούρο, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναμφίβολα, ε, το δημοσιονομικό μέσο το οποίο έχει στη διάθεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα αποτελεί ένα ε, εργαλείο ε, ε, χρήσιμο. Αναφέρομαι βεβαίω στο Ταμείο Αλληλεγγύη. Αλλά είναι αλήθεια ταυτόχρονα ότι μέχρι το 2007, όταν θεωρήσαμε σκόπιμο να αντιμετωπίσουμε τις κριτικές όσον αφορά αυτό το μέσο το δημοσιονομικό ε, ετέθηκε το ζήτημα της ευελιξίας. Είναι σημαντικό λοιπόν η διαχείριση να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία κάθε μέρα ανακύπτουν. Για παράδειγμα, είναι σωστό να, ζητάτε, να ζητείτε ε, σύντομος χρόνος, ε, 10, 10 εβδομάδες από τα κράτη-μέλη να δώσουν ε, στοιχεία ε, και πληροφορίες. Αλλά γιατί δεν δίνονται εξίσου γρήγορα και οι απαντήσεις. Ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε ότι εάν ε, ως προσορισμένες ε, πτυχές είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε την, τη ζημιά και τη βλάβη, αλλά αυτό πρέπει να το συνδέσουμε με τη συγκεκριμένη συγκεκριμένη περιοχή που πλήττεται για να καταλάβουμε ποιε είναι ακριβώ οι ανάγκε του, του πληθυσμού. Ε, ακριβώ γι' αυτό ε, και στη Δημοσιονομική Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο γενικότερα έχουν ακουστεί διάφορε ε, παρατηρήσει. Ε, προ το Συμβούλιο, αλλά το Συμβούλιο δεν φαίνεται να προσέχει αυτέ τι παρατηρήσει. Πρέπει λοιπόν να δούμε την πτυχή τη ευελιξία με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε να, ε, το μέσον αυτό, το Ταμείο Ελληνική, και να είναι όσο το πιο αποτελεσματικό για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία όλο και πιο συχνά θα βρίσκουμε μπροστά μα. Ακριβώ γι' αυτό σα λέω, Επίτροπε, το σημείο 3 και το σημείο 11 του ψηφίσματο να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη. Διότι η πτυχή ευελιξία πρέπει να εξεταστεί όχι ε, ω επιταγή εν λευκό στα κράτη-μέλη, αλλά ε, για να κάνουν ό,τι ε, ε, επιθυμούν, αλλά να, να, να δίδεται μια ευφυή απάντηση προ τι πραγματικέ ανάγκε, έτσι ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο το εργαλείο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Περέγιο. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, πράγματι ε, είναι αδιαφυσβήτητο ότι ε, σημειώθηκε πρόοδο ε, τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώ όμω, παρόλα αυτά, ο νότο τη Ευρώπη καίγεται και καίγεται όλο και περισσότερο. Η δική μα απάντηση λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν μπορεί να είναι άλλο ένα ψήφισμα το οποίο απλά και μόνο να αναφέρει τι μεγάλε ανησυχίε που ε, αισθανόμαστε. Οι πυρκαγιέ στα δάση προξενούνται λόγω συγκεκριμένων αιτιών. Αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί κανεί ότι εντείνονται λόγω των κλιματικών αλλαγών. Και σίγουρο είναι ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να απευθύνει έκκληση με σαφήνεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δράσει σύντομα και να θέσει ε, στη διάθεσή μας όλων όλα τα εργαλεία και τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της. Να λάβουμε υπόψη τα θύματα, τις ζημιές, ε, τις ανάγκες αναδάσωσης, όλα αυτά δεν μπορεί ε, να τεθούν στο περιθώριο στο όνομα ε, μιας γραφειοκρατίας ή των πενιχρών πόρων. Πρέπει να αλλάξουμε στρατηγικές, να κινητοποιήσουμε πόρους και να συντονίσουμε με, όσο τον καλύτερο τρόπο τις, τις ε, πολιτικέ πρόληψης, απαιτώντα πολλέ φορέ και από τα κράτη-μέλη να λάβουν τι ευθύνε του, Να καταλάβουμε όλοι, το, το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο τον νότο τη Ευρώπη. Η αλλαγή του κλίματο δεν αφορά μόνο ορισμένα κράτη, αλλά όλα τα κράτη. Είναι ε, πηγή ανησυχία για όλου. Γι' αυτό ένα από τα βασικά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο άμεσο μέλλον είναι να καταφέρουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση στην επόμενη διάσκεψη Κοπεχάγης να πετύχει συγκεκριμένε δεσμεύσει για τη μείωση, τη δραστική μείωση ε, των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Γιατί ε, τα αέρια αυτά αποτελούν βασική αιτία για τι πυρκαγιέ λόγω και τη αλλαγή του κλίματο. Θα πρέπει λοιπόν να εγκριθεί το ψήφισμα αυτό. Και αυτό αποτελεί συγκεκριμένη πρόκληση για το Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να λάβει τι ευθύνε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλουμε πραγματικά, Επίτροπε, ο νότο τη Ευρώπη να εξακολουθήσει να καίγεται με τον τρόπο αυτό. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Λόπε, δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, ε, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς σε αυτή την πρώτη ολομέλειά μας ε, ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το λυπηρό ε, ζήτημα. Τις φυσικές καταστροφές και πιο συγκεκριμένα τις δασικές πυρκαγιές. Για άλλη μια φορά εκφράζουμε τη λύπη μας για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν μέσα στο θέρος του 2009 και που οδήγησαν και σε απώλεια ανθρώπινης ζωής. 20 θύματα ε, στη χώρα μου και μόνο. Γι' αυτό ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ε, εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μας απέναντι στα δεινά που προξενούν στον άνθρωπο αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Τονίζω τις καταστρεπτικές, καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών στις πληγήσεις περιοχές, στον πληθυσμό, στην φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, στο περιβάλλον, στον τουρισμό, στην περιφέρειά μου 22.000 εκτάρια κάηκαν φέτος το καλοκαίρι. Και το 50% από τις εκτάσεις αυτές ήταν προστατευόμενες λόγω ε, του, ε, του ενδιαφέροντος που προξενούν ως ε, τοπία. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Οι, Ευρωπα... οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν μπορούν άλλη μια φορά να εκφράσουν την αδυναμία τους ως προς την προσφορά λύσεων και βοήθειας προς τις πληγήσιες περιοχές. Πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα και να φροντίσουμε έτσι ώστε να αναδασωθούν οι περιοχές αυτό πιο σύντομα. Πρέπει επίση να δράσουμε στο θέμα τη πρόληψη. Να, ε, να, ε, να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή ε, Ομάδα Πολιτικής Προστασίας. Θα πρέπει να εγκριθούν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να αντισταθμιστούν τα κοινωνικά, να αντισταθμιστεί το κοινωνικό κόστος που συνεπάγονται αυτές οι καταστροφές για τους τοπικούς πληθυσμούς, απώλεια εργασίας κτλ. Δεύτερον, απευθύνω έκκληση στην Ισπανική κυβέρνηση που θα αναλάβει από τον Ιανουάριο του 2010 ε, την Προεδρία. Η Ισπανική κυβέρνηση πρέπει ε, να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων και να μεταφέρει ε, στου υπόλοιπου εταίρου τι ανησυχίε τη. Θα πρέπει μέσα στην ημερήσια διάταξη Ισπανική Προεδρία θα πρέπει να υπάρξει το θέμα τη μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Ταμείου Αλληλεγγύη του Κοινοτικού Ταμείου ελληνική. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών σε επίπεδο πρόληψη, καθώ επίση και σε επίπεδο μοντέλου διαχείριση των δασών, έτσι ώστε να μην ευνοούνται στο μέλλον αυτέ οι τεράστιε πυρκαγιέ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κυρία Μπαλζάνη. Δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως ε, μέλος ε, της ε, ομάδας σοσιαλιστών και αφού άκουσα ε, και τις περασμένες, και, ε, και τις περασμένες ημέρες ε, στην Ιταλία στην, τι έγινε στην Γένοβα, στην περιοχή της Λιγουρίας όπου υπάρχει μακριά παράδοση πυρκαγιών καταλαβαίνετε ότι αισθάνομαι και εγώ ότι επήγει η αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ευρώπη γιατί δυστυχώς αυτές οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο συχνά. Δεν θα έπρεπε όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να παραλαμβάνει το φαινόμενο αυτό και θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθεια έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται αυτές οι κυκλικής φύσεως καταστροφές. Και πιστεύω ότι μόνο ε, η Ευρώπη ενωμένη μπορεί να παρέμβει με αποτελεσματικό τρόπο. Ε, έτσι ώστε να ε, προστατέψουμε αυτές τις, τις, τις περιοχές που αποτελούν κληρονομιά όλων γιατί είναι αλήθεια ότι καίγεται όλο και περισσότερο ο νότος της Ευρώπης. Ε, καταλαβαίνετε όμως ότι όταν καίγεται έστω και ένα μικρό ε, κομμάτι του νότου της Ευρώπης, ολόκληρη η Ευρώπη είναι αυτή που καίγεται και καταστρέφεται. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική πολιτική προστασία των δασών ε, και στον τομέα της πρόληψης. Και εδώ ε, μιλώ ταυτόχρονα και με καταπολέμηση κάθε μορφής κερδοσκοπικής δραστηριότητας που συνδέεται άμεσα ή έμεσα με αυτές τις φυσικές καταστροφές. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να ε, υπάρξει πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους ε, χωρίς γραφειοκρατία έτσι ώστε να μετριάσουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτών των φυσικών καταστροφών, αυτών των καταστροφών. Και αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στο Ταμείο Αλληλεγγύης το οποίο αναμφίβολα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περισσότερη ταχύτητα για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των περιοχών που πλήττονται. Ευχαριστώ κυρία Κροστέτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το 2001 ζητήσαμε ένα μηχανισμό ευρωπαϊκό ε, πολιτικής προστασίας μετά την καταστροφή στις 11 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε ένα ταμείο. Υπήρξε η έκθεση Μπαρνιέ η οποία επέμεινε ότι ήταν αναγκαίο να υπάρξει αλληλεγγύη. Ε, σήμερα η αλληλεγγύη εντάξει λειτουργεί, αλλά θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική. Πιο αποτελεσματική λέω, δηλαδή θα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη ταχύτητα. Υπάρχουν δύο σημεία που πρέπει να αναπτύξουμε. Αντιδραστικότητα πρώτα. Ε, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Όσοι ε, είχαν πρόβλημα με τις πυρκαγιές αυτές, ξέρουν ότι οι διαδικασίες ήταν χρονοβόρες. Ε, πέρασε πολύ χρόνος πραγματικά για την εφαρμογή οποιονδήποτε μέτρων. Ενώ ουσιαστικά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ε, πυρκαγιές πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα. Περισσότερη ευκαμψία. Ευληγησία λοιπόν για την εφαρμογή των μέτρων, διότι ο χρόνος είναι πελίτμος. Πρόληψη τώρα. Δεν μιλάμε αρκετά για την πρόληψη. Δεν μιλάμε αρκετά για την πρόληψη, γιατί είναι θέμα επικουρικότητας. Λέμε λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να αποφασίσουν. Όταν νόμος, αυτές οι πυρκαγιές ε, καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα... το περιβάλλον, φύγουν το πιο πολύτιμο των ανθρώπων, δηλαδή την κληρονομιά τους, το σπίτι τους, όταν, τη γη όταν δυστυχώς ε, χάνονται ανθρώπινες ζωές, ε, λοιπόν δεν μπορούμε να μην έχουμε πρόληψη. Είναι εγκληματικό θα έλεγα, εγκληματική αμέλεια. Θα πρέπει να σταματήσει λοιπόν αυτό. Γι' αυτό όμως χρειαζόμαστε χρηματοδοτικά μέσα. Πρέπει να βρούμε τον βέλτιστο προϋπολογισμό ώστε μέσα στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Ας φροντίσουμε λοιπόν ο προϋπολογισμός μας να λάβει πραγματικά υπόψη όλα αυτά τα θέματα. Χρειαζόμαστε εμείς να έχουμε συγκεκριμένη πολιτική για την αγροτική μας πολιτική και τη δασική μας πολιτική ακόμη. Ε, πρόληψη και πόρους λοιπόν. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε η Ευρώπη του Νότου να μην καίγεται μοιραία. Ευχαριστώ κύριος Αρσένης, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για ακόμη μια χρονιά ο Ευρωπαϊκός Νότος πλήκε δυσβάσταχτα από καταστροφικές πυρκαγιές. Αντίστοιχε μεγάλες πυρκαγιές έλαβαν τόπο στη ΣΥΠΑ και άλλες χώρες του αναπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου Αναφίβολα, η κλιματική αλλαγή απειλεί τα δάση στη Μεσόγειο και σε άλλα κρίσιμα σημεία του πλανήτη. Αλλά και η καταστροφή των δασών τη Μεσογείου καταστρέφει την ικανότητα των φυσικών οικοσυστημάτων να απορροφούν τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα ω φυσικέ αποθήκε. Απαιτούνται ευρωπαϊκέ πολιτικέ πρόληψης και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αλλά και η οικονομική στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρε που, όπω η Ελλάδα αυτή τη χρονιά, αντιμετωπίζουν τι πιο βαριέ επιπτώσει. Αναμφίβολα σε συγκεκριμένε χώρε παρουσιάστηκαν τεράστιε αδυναμίε στο συντονισμό των μηχανισμών δασοπροστασία, τη πολιτική προστασία, αλλά και στη λήψη μέτρων πρόληψη που δεν θα πρέπει ποτέ να επαναληφθούν. Φαίνεται επίση ότι τα δάση που βρίσκονται στη ζώνη τριών ωρών από μεγάλα αστικά κέντρα ή σε τουριστικέ περιοχέ απειλούνται συχνότερα από φωτιέ. Πολλοί νιώθουν ότι μπορούν να έχουν προσωπικά ωφέλη από την καταστροφή των δασών μπορούν να φυτεύουν σπίτια και άλλες κατασκευές πιο γρήγορα από ότι τα κράτη μέλη και τα φυσικά οικοσυστήματα μπορούν να φυτεύουν τα δέντρα στα καμένα. πολλές φορές υπάρχουν εθνικές νομοθεσίες που καλλιεργούν τέτοιες νοοτροπίες και στέλνουν τα λάθος, τα λάθος μηνύματα. μια ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των δασών για την αποκατάσταση των καμένων για τη δάσωση περιοχών ακριβώ στα πλαίσια τη ευρωπαϊκή συμβολή στην ε, αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είναι απολύτω αναγκαία όπω είναι και ένα ευρωπαϊκό συντονισμό των δράσεων πρόληψη αντιμετώπιση πυρκαγιών αποκατάσταση δασών και εδάσεων σε νέων περιοχών. και πρέπει να τα δρομολογήσουμε άμεσα ιδιαίτερα εν ώψη των καθοριστικών για το μέλλον του πλανήτη μα διαπραγματεύσεων στη σύνοδο τη Κοπεχάγης. εκεί θα ζητήσουμε από τι αναπτυσσόμενες χώρες να προστατεύσει τα τροπικά δάση θα θίξουμε το κρίσιμο ζήτημα τη συμβολή τη καταστροφή των δασών στι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου κατά. 20%. πρέπει λοιπόν να είμαστε εμεί αυτοί που θα δώσουμε το παράδειγμα εξασφαλίζοντα την απόλυτη προστασία των απειλούμενων δασών των απειλούμενων δικών μα δασών στην ευρώπη που είναι τα μεσογειακά δάση. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πίπερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η διάσταση των δασικών πυρκαγιών υπερβαίνει όντω τι δυνατότητε των μικρότερων κρατών μελών, ιδιαίτερα σε αυτέ τι περιοχέ που πλήττονται ιδιαίτερα. Γι' αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύη. Καλούμε το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο χωρί εμπόδια, γιατί οι περιφέρειες χρειάζονται κατεπηγόντω τα χρήματα αυτά για την πρόληψη, για την αναοικοδόμηση. Το Ταμείο Αλληλεγγύη σε σύνδεση με διάφορα εφιστάμενα προγράμματα θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει βιώσιμα, αλλά κατά τα άλλα η καταπολέμηση των πυρκαγιών έγκυται στην εθνική αρμοδιότητα. Πιο μεγάλε κυρώσει για τον εμπρισμό, περιορισμός των ε, εκτάσεων για 30 έτη όταν αποδεικνύεται εμπρισμός, γιατί πραγματικά χρειάζεται περισσότερη δράση, αλλά και η Ευρώπη πρέπει να κάνει πιο πολλά πράγματα, κυρίως να συντονιστεί καλύτερα. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες αυτές και χρειάζομαι χρειαζόμαστε και καλύτερου κανονισμού για την διασυνοριακή ανάληψη δράση. Περιμένουμε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς ωστόσο να επισέλθουμε στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, χωρίς να παρεμβούμε στι αρμοδιότητε των εθνικών κρατών μελών. Μπορούμε να διανοηθούμε ευρωπαϊκά μέσα πυρόσβεση, αρκεί πρώτα να έχουμε ε, εξειδανικεύσει αν θέλετε τα εθνικά μέσα. Και νομίζω ότι η συζήτηση για την προστασία από τι ε, καταστροφέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάπω πρόημη. Α κάνουμε πρώτα αυτά που πρέπει να κάνουμε πρώτα. Και αυτό τι είναι ευρωπαϊκή βοήθεια για αυτοβοήθεια. Με το Ταμείο Αλληλεγγύη, με την κατάρτιση και με καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Αγιάλα, ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ελληνική μου ε, και τα συλληπιτήριά μας προς τις οικογένειες των θυμάτων. γιατί είναι αλήθεια ότι κάθε ε, καλοκαίρι δυστυχώς θρυνούμε θύματα. Γι' αυτό και αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία η Ευρώπη τελικά να έχει ένα μέσον στη διάθεσή της, το οποίο είναι αποτελεσματικό. Και ίσως ε, και επειδή εγώ είμαι εμπειρογνώμονα σε θέματα οδική βοήθεια και ασχολούμαι θέματα μεταφορών, ίσω κύριε Επίτροπε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι παρόμοιο με το πρόγραμμα δράση για την ασφάλεια στον τομέα αυτό. Δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένη στρατηγική μέσα ε, και όπου, ε, ε, όπως ακριβώς στον τομέα της οδικής ασφάλειας, θα μπορούσαμε να παρεμβαίνουμε άμεσα και να βοηθήσουμε και τους επαγγελματίες για τις συνθήκες εργασίας, την κατάρτισή τους και κυρίως, και αυτό το πολύ σημαντικό, ευαισθητοποίηση, κουλτούρα πρόληψης. Το καταφέρνουμε σιγά σιγά στα θέματα ασφάλειας στους δρόμους. Γιατί να μην το κάνουμε και στο θέμα των πυρκαγιών. Χαιρόμαστε γιατί βελτιώθηκε ο συντονισμός και η αλληλεγγύη και εδώ νομίζω ότι η Ισπανική κυβέρνηση έστειλε τα απαραίτητα αεροσκάφη ε, και συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια ευαισθητοποίηση ε, των χωρών του Νότου. Αλλά θα πρέπει να μα βοηθήσουν και οι χώρε του Βορρά. Ε, και ακριβώ αυτά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη θα μπορούσαν πραγματικά να οδηγήσουν στη δημιουργία ενό σώματο παρέμβαση θα πρέπει ε, να αντιληφθεί όμω και το Συμβούλιο ε, την προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει και σε επίπεδο προστασία ε, του εδάφου αλλά και σε επίπεδο Ταμείου Αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κύριο Φράγκο, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι και αυτό το καλοκαίρι το μεσογειακό δάσος κάηκε στη Μασαλία, στη Νότιο Κορσική, στην Ιταλία, στην Ισπανία και ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα. 400.000 εκτάρια δάσους γίνανε καπνός. Φοβερές ηλικές ζημίες, πράγματα που δεν διορθώνονται. Η βιοπικιλότητα και οι ανθρώπινες ζωές χαμένες. Επαναλαμβάνεται αυτή η κατάσταση χρόνο με χρόνο. Πολλαπλασιαστικό, πολυ, πολυ, πολλαπλασιαστική επίδραση υπάρχει λόγω της υπερθέρμανσης ε, του πλανήτη και γι' αυτό καλό να συνδέσουμε τις δυνάμεις μας για, την, ε, για τα μέτρα κατά των πυρκαγιών. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει ένα πολύ μεγάλο σχέδιο συνεργασίας προστασίας κατά των πυρκαγιών στη Μεσόγειο. Χαίρομαι για τις υπιστάμενες πρωτοβουλίες και ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Στασικές Πυρκαγιές. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Θα ήθελα όμως να μεταρρυθμιστεί το Ταμείο Αλληλεγγύης ώστε να γίνει ένας μηχανισμός αποτελεσματικός που ανταποκρίνεται στις κρίσεις και θέλω ακόμη να ενισχυθεί η δύναμη προστασίας της Ευρώπης που επινοήθηκε από τον Παρνιέ ήδη το 2006 ώστε να μπορεί να επέμβει στην επικράτεια των 27 κρατών μελών και στο εξωτερικό. Νομίζω ότι ένα από τα κλειδιά επίλυσης του προβλήματος των πυρκαγιών είναι οι γνώσεις και οι καλές πρακτικές για την πρόληψη. Ακόμη θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ε, πρωτοποριακό ρόλο των εθελοντών πυροσβεστών και των επαγγελματιών πυροσβεστών. Ε, στην περιφέρειά μου ήταν καταπληκτική παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η κυρία Ρίτα Κόρολα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ το περασμένο έτος. Ήταν πραγματικά ένα από τα πιο λυπηρά έτη για τις ε, πυρκαγιές. Χάσαμε απίστευτα πολλά εκτάρια δάσους και οι επιπτώσεις δυστυχώς είναι γνωστές σε όλους. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες, για παράδειγμα το ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστούμε σε, για πιο μακριά περίοδο για πυρκαγιές. Γιατί το καλοκαίρι είναι πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες στο Νότο. Αλλά και στην Πορτογαλία είχαμε μεγάλες πυρκαγιές. Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι μόνο στις ε, φυσικές συνθήκες. Διαπιστώθηκε ότι στην Καλιφόρνια οι πυρκαγιές οφείλονται και σε κοινωνικές ε, συνθήκες. Η γεωργία, οι οικισμοί, η καλλιέργεια συγκεκριμένων φυτών η συμπεριφορά των αρχών, όπως για παράδειγμα η απροθυμία επίλυσης και διαλεύκανσης των ε, εγκλημάτων αυτών. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός, αλλά δεν εξηγεί από μόνη της τέτοιες καταστροφές οι οποίες επανέρχονται κάθε χρόνο. Θα πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, γιατί οι μελλοντικέ βασικές πυρκαγιές από μας εξαρτώνται να μην ακολουθήσουμε τις ίδιες κακές πρακτικές στο μέλλον. Thank you. Sari, Asia, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συνδέσω τη φωνή μου με αυτή των παραβερνώντων που υποστήριξαν την ανάγκη πρόληψης. Οπωσδήποτε αυτό στοιχίζει λιγότερο από το να αποκαθιστούμε στη συνέχεια τις ζημίες μετά τις ε, πυρκαγιές. Πρόληψη λοιπόν των πλημμυρών και των πυρκαγιών. Ενεργοποιούμε πόρους. Έχουμε δορυφορική παρακολούθηση. Ε, πρέπει να έχουμε και μηχανισμούς προειδοποίησης. Αυτό εδώ και δεκαετίες έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες όπως η Φινλανδία και στο εθνικό μας πρόγραμμα θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε οι πυροσβέστες να είναι σωστά εξοπλισμένοι για να παρέμβουν εγκαίρως όταν ξεκινούν αυτές οι παρκαγιές. Τώρα, οι πλημμύρες. Οι πλημμύρες είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της μεταβολής του κλίματος. Και εδώ χρειάζεται πρόληψη. Χρειαζόμαστε όμως και συμφωνίες όπως αυτές που προβλέπουμε για την Η πρόληψη λοιπόν σημαίνει ότι μπορούμε να παρέμβουμε εθνικά με τα σωστά μέτρα. Θέλουμε τη σωστή δασική πολιτική, προστασία των δασών, τα δέντρα τα οποία προτιμούμε θα πρέπει να έχουν τη σωστή υγρασία ώστε να μην χάνουν την υγρασία τους το καλοκαίρι και τα λοιπά. και ακόμη πρέπει να αναχαιτίζουμε τις πλημμύρες εγκαίρως με φράγματα ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. Αυτά σημαίνουν ότι η ευθύνη είναι στα χέρια των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναλάβει ε, την ευθύνη στη θέση τους. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει αμέλεια, το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι, ε, παρέχει μάλλον βοήθεια σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης. Βεβαίως όμως θα πρέπει να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα στη δασική πολιτική. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ματόχο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κοιτάξτε, ε, μια φωτιά είναι πάντα μια τραγωδία και για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον και σε οικονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και δυστυχώς ε, είχα την ατυχία ε, να ζήσω πολύ καλά στο νησί Πάλμα στα Κανάρια μια πυρκαγιά. Είμαι πεπισμένος λοιπόν θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα ομόφωνα. Ένα ψήφισμα που είναι πλήρες και που ε, ε, δέχθηκε πολλές συνεισφορές και κυρίως ε, πρώτα απ' όλα υπενθυμίζει τα θύματα και τι φόρο τιμή σε όλου αυτού που καταβάλουν κάθε προσπάθεια και σε θεωρητική βάση για την ε, ε, πυρόσβεση. Τονίζω όμω ταυτόχρονα το πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε την ξηρασία, την απερίμωση ε, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που και είναι εκατοντάδε χιλιάδε εκτάρια το χρόνο. Και τέλο, αναφέρονται και οι αιτίε που, επιβα... που επιδεινώνουν την κατάσταση. Η εγκατάλειψη των αγρών, ε, η εγκατάλειψη των δασών ε, και ε, βεβαίω να τιμωρούνται ε, αυστηρά οι εμπριστέ. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε αποτελεσματικά και με συνέπεια. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί μια στρατηγική αντιμετώπιση των κινδύνων, αποτελεσματική στρατηγική ταυτόχρονα για την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών. Ένα πρωτόκολλο ταυτόχρονα για ενιαία δράση. Αλλά είναι σημαντικέ και οι ενισχύσει για την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, για την αποκατάσταση του παραγωγικού ιστού, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και, την, και των απολειών θέσεων εργασία. Και απαιτείται και συντονισμό. Συντονισμό ανάμεσα στα κοινωτικά μέσα, ε, διαθετικά ταμεία, ε, συντονισμό με το ε, Ταμείο Αλληλεγγύη που βεβαίω ε, πρέπει να το ε, αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τη μεταρρύθμιση του. Και, ένα και το μηχανισμό ε, τον οποίο αναφέραμε για την άμεση ταχεία επέμβαση. Πρέπει να εμβαθύνουμε στην ανάλυση των προβλημάτων αυτών. Και πιστεύω ότι και το ψήφισμα αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο προ την κατεύθυνση κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστούμε. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Φερνάντε. Δύο λεπτά, κύριε Φερνάντε. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο ε, και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, γιατί πραγματικά ήρθε η στιγμή για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και έχουμε την υποχρέωση έτσι ώστε όλοι ε, να συμβάλλουμε στην ε, αντιμετώπιση του ζητήματος και ταυτόχρονα ε, και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη βελτιστοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης έτσι ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άμεσα και να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστροφές. Απαιτούνται λοιπόν αλλαγές και ε, σε επίπεδο δασικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά ευρωπαϊκή δασική πολιτική που να έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τα δάση και να ε, προλαμβάνονται οι πυρκαγιές. Πρέπει να πούμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη, στο δικό μου για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, δεν έχουμε καν ένα κτηματολόγιο με την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε ε, όλους τους ε, ιδιοκτήτες ε, γης, όλους τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων που καίγονται για να προβλέψουμε την αναδάσωση. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αναδάσωσης και ρωτώ το εξή. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνουμε όλες αυτές τις δράσεις στο σχέδιο για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας διότι εάν προωθήσουμε δράσεις ε, που αφορούν τον καθαρισμό των δασών, για παράδειγμα, και ε, το αποτέλεσμα αυτών των δράσεων θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραγωγή ενέργειας μέσω της βιομάζας. Καταλαβαίνετε ότι αν ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, τότε είναι σαφές ότι και θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των δασών, αλλά και ε, θα δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση, πράσινε θέσει απασχόληση, που αυτή τη στιγμή η δημιουργία θέσεων απασχόληση είναι βασικό στόχο τη Ευρώπη. Ο κύριο Βανίστερόι. Δύο λεπτά, ευχαριστώ. Είναι σωστό που σε αυτή την πρώτη μέρα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου συζητάμε τις καταστροφές στην Νότια Ευρώπη και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, που προετοίμασαν ένα καλό ψήφισμα. Ωστόσο, πρόκειται και για θέμα ανθρώπινη επαφή. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στον πολίτη. Το είπαμε και συχνά στην προεκλογική μα εκστρατεία. Και είναι και θέμα αλληλεγγύη. Τώρα έχουμε πυρκαγιέ στην Νότια Ευρώπη. Ποιο ξέρει όμως, μπορεί το χειμώνα να πληχθούν άλλε περιφερειέ τη Ευρώπη από πλημμύρε. Στην Επιτροπή πολλές φορές συζητήσαμε για την βελτίωση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Δεν θέλουμε να ζητήσουμε νέα εργαλεία, θέλουμε τα ήδη υφιστάμενα εργαλεία να καταστούν πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Και κύριε Δήμα, το περίεργο εδώ πέρα είναι το εξή ότι εδώ στο Κοινοβούλιο δηλώσαμε πού θα μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, αλλά το Συμβούλιο μας μπλοκάρει εδώ και δύο χρόνια. Σας ρωτώ λοιπόν, υπάρχει κάποια πρόοδος. Έχετε δίκιο. Έχουμε πρόοδου. για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη, αλλά ο φάκελο τον οποίο ζήτησε ε, το Κοινοβούλιο ε, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Είναι ακόμα στην ατζέντα. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, την, ε, το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Ναι, καλό να έχει η Ευρώπη τα δικά της μέσα, αλλά η μεγάλη ευρεία βάση έγινε σε επίπεδο κράτους μέλους. Και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τη βάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση, αν θέλετε, την αναδιάρθρωση, αυτό δεν πρόκειται για θέμα, δεν είναι θέμα κεντρικής ε, ε, διοίκησης. Θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κράτους μέλους. Και εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης. Να χρησιμοποιηθούν λοιπόν τα αποκεντρωμένα εργαλεία. Αυτό ζητάει το ψήφισμα και αυτό θα υποστηρίξουμε αύριο ένθερμα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κανσιάν. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, ε, κοιτάξτε, είναι σωστό το ε, ψήφισμα το οποίο υπέβαλε το ΕΛΚ με τίτλο Φυσικές καταστροφές. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ορισμένα σημεία τα οποία δεν ε, αναφέρθηκαν σήμερα το απόγευμα ή μάλλον αναφέρθηκαν σήμερα το απόγευμα αλλά δεν ε, περιέχονται στο ψήφισμα. το περασμένο καλοκαίρι, εκτός από τις πυρκαγιές, προξενήθηκαν και άλλες καταστροφές ε, και μάλιστα και το περασμένο Σαββατοκύριακο στο νότο τη Ιταλία. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή, το Βένετο, όπου τον Ιούλιο και τον ε, Ιούλιο αντιμετώπισε ε, πολλά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε στο ψήφισμα και τις άλλες φυσικές καταστροφές και όχι μόνο τις πυρκαγιές. Γιατί οι, οι πλημμύρες, οι καλοκαιρινές, είναι και αυτές καινούργιο φαινόμενο. Και ένα από τα σενάρια τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, ως συνέπεια και αυτό ε, των ε, της αλλαγής του κλίματος και της ε, θέρμανσης, υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιμένουμε λοιπόν στα μέτρα πρόληψης και στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών που θα βοηθήσουν την αποφυγή των γεγονότων αυτών ή τουλάχιστον τον περιορισμό των καταστροφών. και, και βεβαίως να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία επιδεινώνουν τις καταστροφές αυτές. Δεύτερον, επειδή ε, στις περισσότερες ε, περιπτώσεις ε, στι φυσικές καταστροφές υπησέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους υπέτειους τις ευθύνες και να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των κυρώσεων. Τέλος, να πω ότι είναι σωστή αυτή η δημιουργία της αυτόνομης δύναμης επέμβασης και ε, η μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Θα πρέπει ταυτόχρονα όμως να διευρύνουμε την επέμβαση και σε άλλες καταστροφές, να ε, αυξήσουμε ε, τα κονδύλια τα οποία θα διατηθούν για το σκοπό αυτό, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει περισσότερο συντονισμός και περισσότερη ευελιξία. Θέματα, θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος Μάουρο. Ευχαριστώ. Κύριος Καντσιάν ο τελευταίος ομιλητής στο κατάλογο. Και τώρα θα ακολουθήσουμε την διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μαγκίνες βλέπω ότι ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τη συζήτηση αυτή από το γραφείο μου και προφανώς στην Ιρλανδία δεν έχουμε ευτυχώς ε, τόσο έντονα προβλήματα όσο στην Νότια Ευρώπη. Και δύο πράγματα με εντυπωσίασαν. Καταρχάς ότι μιλάμε εδώ στο Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά που επηρεάζουν κυρίως τι δικέ μας χώρες. Και εμείς στην Ιρλανδία συζητάμε για το δημοψήφισμα και μιλάμε για την αλληλεγγύη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτή την συνήθεια θα πρέπει να την ε, σπάσουμε. Θα πρέπει να μιλάμε όλοι για θέματα που αφορούν άλλα κράτη-μέλη. Προκειμένου να υπάρχει όντως μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των βουλευτών του Κοινοβουλίου αναφορικά με τις ανησυχίες των ε, πολιτών για παράδειγμα θα ήθελα και άλλοι να ανησυχήσουν και να μιλήσουν για τις ανησυχίες των πολιτών στην Ιρλανδία. Όλα αυτά θα μας βοηθούσε να προωθήσουμε την ιδέα ότι η Ευρώπη λειτουργεί για όλους και ότι δεν κοιτάμε απλά τα δικά μας, ε, τα, το δικού μας οίκου. Αυτό αποτελεί μια αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πραγματικά ε, μας, ε, επιζημιώ, μας, δεν μας ωφελεί στη συζήτηση για, την, ε, το Ιρλανδικό δημοψήφισμα. Άρα θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στους εμπριστές. Και τέλος, όντως, να απελευθερώσουμε τα ταμεία αλληλεγγύης για όσους τα χρειάζονται. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Λόπες. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά. Ε, η πρώτη μου λοιπόν εκλογή στις, ε, τον Ιούνιο. Αλλά ήδη ε, για μένα είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό ανακύπτει κάθε Σεπτέμβριο μετά από το κύμα των πυρκαγιών ε, που ξεσπούν ε, το καλοκαίρι, κυρίως στον νότο της Ευρώπης, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Αναφέρθηκε η, καταστροφική πυρκαγιά στο νησί Πάλμα, στα Κανάρια, αυτόνομη περιφέρεια της Ισπανίας στην οποία ε, το φαινόμενο αυτό ε, παρουσιάζεται ε, επανειλημμένα. Ναι, είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο στον νότο της Ευρώπης, αλλά αυτό αποτελεί θαυμάσια ευκαιρία για να συσφίξουμε τους δεσμούς μας όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τι σημαίνει Ευρώπη? Προστιθέμενη αξία λοιπόν, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο πρόληψης, επίπεδο συντονισμού των θεσμών, Επιτροπή, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Προσθέμενη αξία ευρωπαϊκή και όσον αφορά τι απαντήσει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε από τη θεωρία στα, ε, στην πράξη. Ε, Βεβαίω το Ταμείο Αλληλεγγύη θα πρέπει να το καταστήσουμε περισσότερο ευέλικτο και ε, να ε, αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα που εκκρεμεί την ευρωπαϊκή δύναμη παρέμβαση, γιατί αυτό θα αποτελέσει την πραγματική προσθέμενη αξία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι και λόγω τη ε, αλλαγή του κλίματο. Σα ευχαριστώ, κυρία Φιγκουρέιδο. Ένα λεπτό. Εκτός μικροφώνου. Οι πυρκαγιές λοιπόν στα δάση αποτελούν ε, μια πραγματική πληγή ε, για τις χώρες του Νότου κάθε χρόνο. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιστοιχούν τρέψουμε αυτή την τάση. Γιατί ε, πρόκειται ε, για την πολιτιστική μας κληρονομιά, για τα ζώα μας, τα φυτά μας, τα δάση μας. Ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ, έχουν τρομερές, τρομερά καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε υπόψη συνδυασμό με την έξοδο από την Ήπεθρο, αποτέλεσμα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Και εγώ πιστεύω ότι πραγματικά ε, η γεωργία και οι γεωργικές δραστηριότητες θα πρέπει να διαφοροποιηθούν πολύ περισσότερο. Να βοηθήσουμε τους μικρούς ε, ιδιοκτήτες των, ε, τους ιδιοκτήτες των μικρών εκμεταλλεύσεων, τους αρχηγούς των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, τους νέους έτσι ώστε να μην φεύγουν από την Ήπεθρο. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, με την πρόληψη και θα καταπολεμήσουμε αυτή την πληγή που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Ε, σας ευχαριστώ. Η επόμενη μιλήτρια για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι ο Επίτροπος Δήμας σχολίασε αυτή την υπόθεση και υποχωράμισε την σπουδαιότητα των ενισχύσεων πέραν των συνόρων της πύρους μας. Μέσα στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα μπορούσαμε να προβλέψουμε εκτός από την οικολογική προστασία της Μεσογείου και αυτή την επίγουσα ενίσχυση σε περίπτωση ε, πυρκαγιών. Αναπτύσσοντας την πραγματογνωμοσύνη μας ε, σε αυτόν τον τομέα και ε, μοιράζοντας τις γνώσεις μας μεταξύ των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο σας. Ο κύριος Λουάν είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φέτος το καλοκαίρι η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα είχαν να αντιμετωπίσουν φοβερές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα οι πυρκαγιές έθεσαν σε κίνδυνο 21.000 εκτάρια, κατέστρεψαν σπίτια, οικισμούς. Χρειάζεται λοιπόν να συντονιστούμε. Η Γαλλία και η Κύπρος και η Ισπανία έστειλαν αεροσκάφη για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Η ευρωπαϊκή στρατηγική μοιάζει να ήταν σωστή ήταν χρήσιμη. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπωσδήποτε μπορεί να παρέμβει σε αυτού του είδους της καταστάσεις αναλαμβάνοντας κάποιες λαπάνες ώστε να αποκατασταθεί η υποδομή, να προστατευθούν άμεσα οι άνθρωποι, να μπορέσουν να τους δοθεί μια προσωρινή κατοικία κτλ. Χρειαζόμαστε όμως λιγότερη γραφή φιοκρατία και επιμένω για να μπορούμε να έχουμε πραγματική πρόσβαση σε αυτό το τομείο. Στη χώρα μου, πέρσι τον Ιούλιο, υπήρξαν φυσικές καταστροφές φοβερές. Φέτος, είμαστε στο Σεπτέμβριο 2009 και ακόμη τα ε, ε, σχετικά κονδύλια δεν έχουν δοθεί στη ρουμανική κυβέρνηση. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μια πραγματική δασική πολιτική, μια στρατηγική παρέμβαση. Σε ευχαριστώ. Τέλος, το λόγο έχει ο κύριος Δήμας για να συνοψίσει και να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις τους, πάρα πολύ βοηθητικές ε, στην απόψινή συζήτηση και τις πολύ καλές ιδέες τις οποίες πρότειναν οι καταστάσει έκτακτης ανάγκης συχνά συνεπάγονται υψηλό ανθρώπινο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής όπως τονίστηκε από πολλού συναδέλφου, πιθανότατα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες καταστροφές όχι μόνο ε, δασικέ πυρκαγιέ, οι οποίε δεν θα περιορίζεται μόνο στο νότιο της Ευρώπης αλλά και στην κεντρική Ευρώπη και ακόμη και στο βορρά της Ευρώπης αλλά και άλλου είδους καταστροφές όπως είναι ε, οι πλημμύρες. Χρειάζεται επομένω να ενισχύσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τα ευρωπαϊκά μέσα διαχείριση των καταστροφών, τα οποία έχουν πλέον σαφές αποδείξει την προστιθέμενη αξία τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, που μας υπενθύμησαν ότι η κοινότητα οφείλει να βελτιώσει όχι μόνο την ικανότητα ανταπόκρισης στις φυσικές καταστροφές αλλά επίσης και τη δυνατότητα πρόληψής τους. Αυτό τονίστηκε από πολλούς ομιλητές απόψε. Και εδώ θα πρέπει να σας θυμίσω ότι το Φεβρουάριο η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση, παρουσίασε ανακοίνωση σχετικά με την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και των καταστροφών ε, που οφείλονται στους ανθρώπους στην οποία διατύπωσε ορισμένες προτάσεις. Αναμένουμε τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ε, και πιστεύω ότι το, αυτό το κοινοβούλιο, το νέο κοινοβούλιο, δεν θα καθυστερήσει στην απάντησή του. Περιμένουμε από το Φεβρουάριο. Πιστεύουμε ότι θα μας δώσουν το πολιτικό κίνητρο μαζί με την ε, τη resolution που, το ψήφισμα το οποίο θα ε, ψηφιστεί ε, στην επόμενη για να προωθήσουμε τις σχετικές διεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι γιατί πολλοί ανεφέρθησαν, κυρία Ποδηματά ξεκίνησε αλλά και πολλοί άλλοι μίλησαν για το θέμα της κλιματικής αλλαγής ε, και της αναγκαίας προσαρμογής η οποία χρειάζεται ε, και την ε, προτινόμενη αναθεώρηση της κοινοτικής στρατηγικής για τα δάση με στόχο να αντιμετωπιστούν πτυχές οι οποίες είναι συναφές με το κλίμα. Θα αποτελέσει και αυτή ευκαιρία για να εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές. Πρέπει εδώ να σας πω ότι αυτή η ανακοίνωση την οποία έκανε η Επιτροπή είναι πολύ σημαντική, όπως πολύ σημαντική είναι και η ανακοίνωση την οποία κάναμε την περασμένη εβδομάδα για την χρηματοδότηση ε, των κλιματικών, της συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές που αναμένουμε στην Κοπενχάγη, μεταξύ των οποίων και ένα μεγάλο ε, ε, ποσό θα πάει για την χρηματοδότηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα έργα εκείνα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουν αυτές οι χώρες οι οποίες υφίστανται τις ε, επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές χωρίς να έχουν συντελέσει στη δημιουργία του φαινομένου του ε, θερμοκηπίου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις, τις επιπτώσεις. Και μάλιστα έχω προτείνει όχι απλώς να περιμένουμε το 2013 για να αρχίσουμε αυτή τη δράση, αλλά να ξεκινήσουμε αμέσως από το 2010 και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είτε στις 17 αυτού του μήνα είτε ε, τον Οκτώβριο θα συμφωνήσει ώστε να δοθούν χρήματα ε, για, την, ε, για να ξεκινήσουν τα έργα αμέσως ώστε και οι χώρες αυτές να δούνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες εννοούν αυτά τα οποία προτείνουν και τα οποία διακηρύσσουν. Πολλά επίσης άκουσα και πολύ σημαντικά και ε, μπορώ να πω ότι όλα είναι σωστά σχετικά με το ρόλο των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων. Ο κοινοτικό κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη προσφέρουν τη δυνατότητα στήριξη εθνικών μέτρων πρόληψη η επιτροπή θα χρησιμοποιήσει επίσης τις δυνατότητες που προσφέρονται από το κοινοτικό ταμείο αλληλεγγύης ώστε να υποβοηθήσει τις προσπάθειες ε, αποκατάστασης στα κράτη μέλη. εδώ πρέπει να πω γιατί άκουσα για την, ε, το ότι πρέπει η παρέμβαση από, ε, από, την επιτροπή να είναι άμεση. Και έχουμε δύο θέματα δεν, ήταν, δεν έγινε πλήρης διευκρίνηση σε ποιο από τα δύο είναι ένα για την, κινητοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και το άλλο είναι για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ως προς το θέμα της ε, κινητοποίησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας μπορώ να σας πω ότι οι κινητοποίηση είναι άμεσος, σε real time, αμέσως. Στις φωτιές, χάρη πρόσφατα, θα σας αναφέρω το παράδειγμα της Ελλάδος, σε μία ώρα αφότου μας ειδοποίησε, μας υπευλήθη το επίσημο αίτημα από τις, την ελληνική κυβέρνηση ιταλικά αεροπλάνα σε μία ώρα είχαν ξεκινήσει ε, για να βρίσκονται ε, και να επιχειρήσουν ε, την επόμενη μέρα. Επομένως οι κινητοποίηση είναι άμεση. Σας είπα δε και στην, στην πρώτη μου ομιλία ότι ήμασταν οι πρώτοι στις περιπτώσεις του τσουνάμι και της Κατρίνα οι οποίοι στείλαμε ειδικού στους χώρους της, των καταστροφών και ε, οι έπαινοι τους οποίους έχουμε δεχθεί για την δραστηριότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας είναι πάρα πολλοί οι οποίοι επιβεβαιώνουν και το έργο το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αλλά και τις δυνατότητες τις οποίες έχει εφόσον έχει αρμοδιότητες και τα μέσα κυρίως χρηματικά να μπορέσει να επεκτείνει ε, το έργο της επωφελία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, ως προς το Ταμείο Αλληλεγγύης, ε, άκουσα και σωστό είναι ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ε, ε, ευελιξία και πράγματι και χρειάζεται το, να, μπορεί να όσο το δυνατόν γρήγορα γιατί ακριβώς στη φιλοσοφία του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι η κάλυψη των αναγκών, ημέρους των αναγκών για των επιγουσών αναγκών οι οποίες προκλήθησαν από τις καταστροφές. επομένως λογικό είναι και η επιτροπή να πρέπει να δρά αμέσως αλλά και τα κράτη μέλη είτε οι κεντρικές διοικήσεις τους είτε οι περιφερειακές ε, διοικήσεις τους ε, να ε, προχωρούν στην ε, σε, άμεσες ενέργειες ώστε και τα χρήματα να εκταμιεύονται. Εξάλλου υπάρχει και ο όρος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης ότι μέσα σε ένα χρόνο από την εκταμίευση πρέπει να έχουν γίνει τα έργα. Λογικό είναι. Αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη ε, ε, ευελιξία. Κλείνοντας, επειδή λυπάμαι που δεν έχω περισσότερο χρόνο να απαντήσω στα πολύ συγκεκριμένα θέματα, να πω μόνο πριν το ξεχάσω για το γιατί άκουσα αρκετούς ομιλητές να αναφέρονται στα ε, σχέδια ανάκαμψης, τα προγράμματα οικονομικής ανάκαμψης. Πράγματι, είναι πολύ καλή ιδέα. Γιατί το να έχουμε, ε, να συμπεριλάβουμε έργα για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, οι οποίες περίπου μπορούν να προβλεφθούν ότι θα συμβούν και τον άλλο χρόνο. Βλέπουμε, ε, λέχθη προηγουμένως, κάθε χρόνο τα συζητάμε τα θέματα αυτά. έχει πολλαπλά ωφέλη και ωφέλη γιατί θα προκαλέσουν οικονομική δραστηριότητα και περισσότερες θέσεις απασχόλησης αλλά επίσης γιατί θα αποτρέψουν τις ζημιές εκατομμυρίων ε, ε, ευρώ ε, για την αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν. επομένως είναι επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν πολλαπλά και βεβαίως θα αποτρέψουν και, την, το ανθρώπινο κόστος των, από τις καταστροφές. Κλείνοντα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ενώ ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών ή άλλων καταστροφών όπως είναι πυρκαγιές σεισμοί ακόμη και στρατιωτικές επεμβάσεις γιατί ο μηχανισμός ε, πολιτικής προστασίας ευρωπαϊκής ε, ένωσης έχει επέμβει και για πλημμύρες και για ε, σεισμούς και για δασικέ πυρκαγιές αλλά και για μετακινήσεις πληθυσμών παραδείγματος μετά τη σύγκρουση στο λίβανο με μεγάλη επιτυχία. πολύ, ε, ε, βοηθήσαμε πάρα πολύ στο, στο θέμα αυτό. Ε, ε βεβαίως ενώ οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν ποτέ να εξαλειφθούν εντελώ εν τούτης μπορούν να μειωθούν μέσα από τη συνεργασία μα και την καλύτερη συλλογική ανταπόκριση σε τέτοιου είδου καταστροφέ. η επιτροπή δεσμεύεται να ενισχύσει την κοινοτική συμβολή στην πρόληψη την ετοιμότητα την ανταπόκριση και την αποκατάσταση καταστροφών ώστε να προστατεύσει του πολίτε και το περιβάλλον. επιθυμώ και πάλι να ευχαριστήσω το κοινοβούλιο που στηρίζει ένθερμα την ανάγκη βελτίωση τη διαχείριση των καταστροφών προ όφελο όλων των ευρωπαίων πολιτών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε γιατί ήρθατε σήμερα και γιατί μας ε, δώσατε αυτές τις απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έληξε η συζήτηση για το θέμα αυτό. συμφορία θα γίνει την Τετάρτη. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η δήλωση της Επιτροπής για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Νότιο Κορέα και βεβαίως ε, ε, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τον αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Σας ε, παρακαλώ, Λέδη Άστο, να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε ένα μεγάλο δυναμικό νέων εξαγωγικών δυνατοτήτων εμφανίζεται στις ασιατικές αγορές που έχουν βεβαίως μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό αλλά και εμπόδια